Ενημερώνω ότι η γραπτή δήλευση 0068 του 2010 από τους Μποκ Μπρεπόνς, Σίλβιο Μπουσόη, Γιώ Λάιενεν και Πέτερλε για την καταπολέμηση του καρκίνου του ορθού στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αριθμό υπογραφών ανώτερο της πλειοψηφίας των Ευρωβουλευτών του Κοινοβουλίου και επομένως θα διαβιβαστεί και θα δημοσιευτεί στα κείμενα που εγκρίθηκαν ε, στη συγκεκριμένη Σύνοδο της Ολομέλειας. Θέλει το λόγο ο κύριος Ποκ. Ε, είναι στο ημικύκλιο. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι ε, γνωρίζω ότι όλοι θέλουν να ψηφίσουν βέβαια, αλλά θα ήθελα εκ μέρου όλων των συνυπογραφών των Μπούσολ, Μπρέπελ, ε, Γιολάινεν, του υποφαινομένου. Να σας ευχαριστήσω που μας υποστηρίζετε στην πρόταση κατά του καρκίνου. Έρχεται η στιγμή εγκαίρως να προχωρήσει το θέμα αυτό και ήθελα να επισημάνω ότι ε, δεν είναι μια μεμονωμένη κίνηση αυτή, αλλά αντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια απευθυνόμενη στα κράτη-μέλη. Σας ευχαριστώ. Η 0065 του 2010 που υποβλήθηκε από τους συναδέλφους Βιντάλ, Κουάντρας, Σόντεργαν, Σίβενσον και άλλους